der präsident! Επανάληψη τη Συνόδο. Καλημέρα σα και πάλι. Να σα ε, ανακοινώσω τα αποτελέσματα τη δεύτερη ψηφοφορίας. Θα τα βρείτε και, στε, και στους πίνακες και θα εκτυπωθούν και θα τα βρείτε και στο homepage. Θα σας, ε, δεν θα σας διαβάσω τα μεμονωμένα αποτελέσματα. Δεύτερη τροπολογία για το ψήφισμα για την ε, διαμαρτυρία κατά του ρατσισμού μετά τον θάνατο του Φλόιτ. Και, και τα τέσσερα τμήματα εγκρίθηκαν. Η 42 τροπολογία εγκρίθηκε, η 3 τροπολογία εγκρίθηκε, τροπολογία 16 απορρίφθηκε. Τροπολογία 443 εγκρίνονται. Τροπολογία 58 απορρίπτεται. Τάφ σε δύο τμήματα αρχικού κειμένου. Σε τι τμήματα λοιπόν. Και τα δύο εγκρίνονται. Ε, τροπολογία 9 απορρίπτεται. Τροπολογία 59 εγκρίνεται. Recital U. Αρχικού κειμένου α, καταπίπτει, το οποίο ήταν σε δύο πτήματα. Η 60 τροπολογία απορρίπτεται, 17 απορρίπτεται, 34 απορρίπτεται, 5 απορρίπτεται, 18 απορρίπτεται και 19 απορρίπτεται. το θέμα της ε, εθνικής ε, ασφάλειας για την Κίνα, Χογκόν και ανάγκη για μέτρα αυτονομίας. Παράγραφος 1 αρχικού κειμένου εγκρίνεται. Τροπολογία 8 απορρίπτεται, τροπολογία 9 απορρίπτεται, τροπολογία 10 απορρίπτεται, τροπολογία 11 απορρίπτεται, 12 απορρίπτεται. Παράγραφος 6 αρχικού κειμένου σε... και τα τρία τμήματα εγκρίνονται. Τροπολογία 6 απορρίπτεται, 13D Επίση απορρίπτεται παράγραφος 13 παράγραφο 12 αρχικού κειμένου εγκρίνεται, 12, 13 αρχικού κειμένου εγκρίνεται, 15 αρχικού κειμένου εγκρίνεται, 22 αρχικού κειμένου και τα δύο τμήματα εγκρίνονται, τροπολογία 1 απορρίπτεται, 2 απορρίπτεται, 3 απορρίπτεται, 4 απορρίπτεται, 5 απορρίπτεται, 7 απορρίπτεται. Και περνάμε στο θέμα της Ανατολικής Ιατρικής Σχέσης. Πριν από τη Σύνοδο του 2020, η τροπολογία 1 9 ψηφίστηκαν ε, ομαδικά, απορρίφθηκαν. Παράγραφος 1, σημείο W, αρχικού κειμένου, εγκρίνεται. Το κείμενο για την κατάσταση του Σέγγεν μετά την ξέσπασμα 19 Έχουμε ψηφοφορία συνολικά 1 έως 3 τροπολογίες, 5, 6 και 10 έως 11 απορρίπτονται όλες αυτές. Η ε, τροπολογία 7 απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παραγράφος 7 και τα δύο τμήματα εγκρίνονται. Τροπολογία 8 απορρίπτεται. Η 9 απορρίπτεται επίσης αρχικού κειμένου. Παράγραφος 13 και τα δύο τμήματα εγκρίνονται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 15 και τα δύο τμήματα εγκρίνονται. Παράγραφος 16 αρχικού κειμένου εγκρίνεται. Παράγραφος 17 αρχικού κειμένου εγκρίνεται. λογική σκέψη Β και τα δύο τμήματα εγκρίνονται. Ε, σκέψη Ε εγκρίνεται. Τροπολογία 4 απορρίπτεται. Τροπολογίε. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο, να κοιτάξουμε το κείμενο για την Ευρωπαϊκή Προστασία των Εποχιακών και Διασυνοριακών Εργαζομένων σε ό,τι αφορά το ξέσπασμα του COVID-19. Τροπολογίε 3, 6 και 10 απορρίπτονται. Τροπολογία 14 απορρίπτεται. Τροπολογία 12 εγκρίνεται. Τροπολογία 15 απορρίπτεται. Τροπολογία 16 απορρίπτεται. Παραγραφός 4 αρχικού κειμένου εγκρίνεται. Τροπολογία 4 και 7 απορρίπτονται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 14 εγκρίνεται, 13 τροπολογία απορρίπτεται, τροπολογία 8 εγκρίνεται και καταπίπτει το αρχικό κείμενο της παραγράφου 19 και τα δύο τμήματα. Παράγραφος 20 αρχικού κειμένου εγκρίνεται. Παράγραφος 23 τροπολογία 1. Σημείο 1 εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα όμως απορρίπτεται. Τροπολογία 11 εγκρίνεται και οι ταυτόσημες 2 και 5 και 9 εγκρίνονται. Τροπολογία, συγγνώμη, ε, λογική σκέψη ο, ο μικρόν ε, εγκρίνεται. Π επίσης εγκρίνεται το αρχικό κειμένο. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του δεύτερου γύρου και περνάμε στο δεύτερο, τρίτο γύρο ψηφοφοριών που ξεκινάει από τώρα μέχρι τις 7.19 η ώρα. Θα ισχύσουν οι ίδιε διαδικασίε και ξεκινάει λοιπόν έτσι ούτως ο τρίτος γύρος ψηφοφορίας. Έχετε μέχρι τις 7 να ψηφίσετε. Τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου θα ανακοινωθούν από την Ολομέλεια στις 9.30 το βράδυ. Λίγη τη συνεδρίαση.